Dear ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Welcome Καλώς ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Σημείο 1 είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Να σας ενημερώσω για κάτι. Το σημείο 8 θα εξεταστεί μετά από το σημείο 26, τα σημεία 14. 23 αλλά και 25 αναβάλλονται και το σημείο 30 θα συζητηθεί μετά από το σημείο 12. Έχετε αντιρρήσεις? Δεν βλέπω. Άρα η ημερήσια διάταξη θεωρείται ως εγκεκριμένη. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το εργαστήριό μας για την αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 θα λάβει χώρα αύριο από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 6.30 το απόγευμα εντάφθα σε αυτή την αίθουσα. Αυτή είναι η μόνη ανακοίνωση. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και αν δεν παραληφθούν ενστάσεις μέχρι το τέλος συνεδριάσεως, τα πρακτικά τη συνεδριά τη 26 Σεπτεμβρίου του 2016 θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Πάμε στο σημείο 4. Συζητούμε τις τροπολογίες που αφορούν τους κανόνες του αστικού δικαίου για τη ρομποτική και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια που είναι η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι σαν προθεσμία για μετάφραση των τροπολογιών και ήταν μέχρι τις 11 σήμερα δεν είχα χρόνο να τις δω τις τροπολογίες μπορώ να σας πω ότι 386 τροπολογίες υπευλήθησαν στα και έχουν έξι, έξι επιτροπές υπάρχουν που γνωμοδοτούν επί της εκθέσεως. Για την ώρα η ΙΜΚΟ, ΙΤΡΕ και ΕΝΒΗ, τρεις επιτροπές έχουν υθετήσει γνωμοδοτήσεις και τρεις άλλες επιτροπές, ΕΜΠ, ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ, θα ψηφίσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Όλες οι επιτροπές όμως, πρέπει να σας το πω αυτό, έκαναν πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατο να μας στηρίξουν. Θέλουμε μια σφαιρική εικόνα των μελλοντικών εξελίξεων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά θα είναι πρόβλημα να αποφύγουμε τις επαναλήψεις, διότι σχεδόν κάθε επιτροπή έχει υπερβάλει εαυτόν και έχει υπερβάλει κάπως τα όρια της όσον αφορά δεξιότητες, προστασία των δεδομένων, ε, προσόντα και αυτά τα στοιχεία αναφέρονται σχεδόν σε κάθε γνωμοδότηση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εισηγητές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των επαναλήψεων. Έριξα μια ματιά στις τροπολογίες που υπευλήθησαν στη δική μας ε, Επιτροπή. Φαίνεται ότι τα βασικά προβλήματα που πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερώς είναι οι ευθύνε, ασφάλιση, δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη και είναι διχασμένες οι απόψεις λόγω των θεμάτων. Εγώ επέβαλα κάποιες τροπολογίες να σας πω κάποια πράγματα για αυτές. Θα τονίσω την αρχή της διαφάνειας. Κυρίως πρέπει να είναι δυνατόν η τεχνητή νοημοσύνη να έχει τέτοια μορφή που να είναι κατανοητή από τον άνθρωπο, από τον ανθρώπινο εγκέφαλο διότι φοβάται ο κόσμος για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ε, πολύ συχνά δεν κατανοούμε τους αλγορίθμους που δημιουργούν τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να προβλέπετε υποχρέωση για εκείνους που ετοιμάζουν το λογισμικό με εύλητο τρόπο να εξηγούν ακριβώς περί τίνος πρόκειται ο αλγόριθμος ε, και πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Επέβαλα μια τροπολογία λέω ότι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για τη ρομποτική θα μπορούσε να είναι αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση της διαφάνειας. Θα δίνει ένα σήμα περί διαφανείας. Θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ευθύνες, τις ενδεδειγμένες, το πλαίσιο των ευθυνών ε, και για τη διαχείριση του κινδύνου επίσης, ποια προσέγγιση θα ακολουθήσουμε. Στις ακροάσεις ακούσαμε πολλά περί προσεγγίσεως διαχειρίσεως του κινδύνου και θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη αξιολόγηση αυτού μέχρι να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να ισχύει η αυστηρό καθεστώς για τις ευθύνε ή η μέθοδος διαχείρισης του κινδύνου. Οι ευθύνε του καθεστώς ευθυνών απαιτούν έγκριση και απόδειξη ότι ε, υπήρξαν ζημίες και σχέση ε, αιτίου και αποτελέσματος. Δηλαδή ότι δεν λειτουργήσε σωστά το ρομπότ και προξένησε ζημίες. Η προσέγγιση διαχειρίσεως του κινδύνου δεν εστιάζεται επί εκείνου που έδρασε ένα μελία αλλά επί εκείνου που είναι υπεύθυνο σε κάποιες περιστάσεις να λαχιστοποιεί τον κίνδυνο και να αντιμετωπίζει τις αρνητικές συνέπειες. Αυτές ήταν οι τροπολογίες που με απασχόλησαν τα επόμενα βήματα. Θα γίνει συνεδρίαση των σκιωδών την 5η, 10 ε, Νοεμβρίου. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει προγραμματιστεί για την 28 Νοεμβρίου και ελπίζουμε να ψηφίσουμε στην Σύνοδο του Ιανουαρίου στην Ολομέλεια. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μαρίνιο Επίντου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφο την κυρία Ντελβό. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω και κάποιες αμφιβολίες. Αμφιβολίες όσον αφορά τα ρομπότ και τη ρομποτική τεχνολογία και όλο το θέμα. Από όταν είδα την ταινία του Κιούμπρικ 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Από τότε και εγώ έχω αμφιβολίες Είδαμε εκεί ότι ένα ρομπότ, ένας υπολογιστής, εξολοθρεύει τους ανθρώπους και το κάνει από ματοδοξία. Ε, εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι αυτή η ουτοπική πραγματικότητα που δημιούργησε ο Κιούμπρικ στον κινηματογράφο, αλλά το θέμα της ρομποτοποίησης της παραγωγής, της βιομηχανικής παραγωγής, της παροχής των υπηρεσιών κλπ. Κατά το παρελθόν ε, είχαν επαναστατήσει εργαζόμενοι κατά της βιομηχανικής επανάστασης και της ε, χρήσης μηχανών για την κλωστεφαντουργία. Τώρα όμως πρέπει να πούμε ότι το ρομπότ δεν θα αμείβεται ποτέ, άρα δεν θα είναι ποτέ καταναλωτή το ρομπότ. Άρα θα είναι απο... απειλή για την οικονομία της αγοράς το ρομπότ, τα ρομπότ. Διότι Πάντα στην οικονομία της αγοράς έχουμε το πρόβλημα της υπερπαραγωγής. Δηλαδή αυτό οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφά τα παραγόμενα. Αν ροποτοποιήσουμε λοιπόν την παραγωγή θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Δεν θα απορροφώνται τα παραγόμενα προϊόντα. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει αναλυθεί στην προσέγγιση του θέματος. Όσο με αφορά με προβληματίζει αυτό. Ανησυχώ τα μάλα. θα είναι δύσκολο να μπορούμε να συμμετάσχουμε σωστά στις εξελίξεις στο μέλλον. Ανησυχώ όμως, σας το λέω, ανησυχώ από αυτό που σας είπα. Δηλαδή, η ρομποτοποίηση ε, δημιουργεί κάποιο ενδιαφέρον, είναι κάτι ελκυστικό, είναι κάτι ενδιαφέρον. Όμως, αν ρομποτοποιηθεί πλήρω η βιομηχανική παραγωγή, η μέθοδη υπολογισμών κλπ. κλπ. Διερωτώ με σε ποιο βαθμό αυτή η ρομποτοποίηση θα κάνει τον άνθρωπο να πάει σε μια θέση ε, υποδέστερη. Θα είναι μια κρίση όπου το βασικό θύμα θα είναι ο άνθρωπος. Ευχαριστώ. Δεν ε, βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος ε, το λόγο. Ο κύριος Άντερσον έχει το λόγο. Πρώτος εσείς, κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ. Δεν διάβασα ακόμα όλες τις τροπολογίες. Συνέταξα 25 από αυτές. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά καλές. Δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες εδώ. Θέλω να αναφέρω τα στοιχεία των σημαντικότερων τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα όταν κάτι πάει στραβά. Θα ήταν χρησιμότατο να έχουμε πρόσβαση στον κώδικα πηγής του λογισμικού. Να δούμε τι πήγε στραβά για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων που δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε αυτό το σημείο, στην πηγή του λογισμικού. Είναι να δυσχεραίνεται πολύ η ανάλυση του κώδικα πηγής του λογισμικού. Έχω και μία τροπολογία για ενδεχόμενους μακροπρόθεσμους κινδύνους. Λόγω της δημιουργίας υπολογιστών που είναι ευφιέστεροι των ανθρώπων. Δεν γνωρίζουμε αν είναι τεχνολογικά εφικτό τώρα, αλλά θα μπορούσε να συμβεί και θα ήταν πολύ καλό αν η έρευνα περί της αντιμετωπίσεως τέτοιων προβλημάτων να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αν προκύψουν. Έχουμε λοιπόν μια σχετική τροπολογία. Άκουσα κάποιες παράξενες επικρίσεις που αφορούσαν την έκθεση. Σύμφωνα με αυτές, μάλλον εσφαλμένα, ότι η έκθεση θέλει να δώσει ανθρώπινα δικαιώματα στα ρομπότ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό μας είπε και η συγκίτρια. Αλλά έχουμε σημείο στην έκθεση περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η έκθεση αναφέρεται σε πνευματικά δικαιώματα για δημιουργήματα της τεχνητής εφίας συγγραφή άρθρων Φερρυπίν. Ακόμα και σήμερα η συγγραφή άρθρων μπορεί να πραγματοποιηθεί από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα για τα πνευματικά δικαιώματα, υποτίθεται ότι αυτό τα πνευματικά δικαιώματα αντικατοστρίζουν την προσωπικότητα του συγγραφέα. Και δεν πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο όπου είναι εύλογο να δώσουμε πνευματικά δικαιώματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε σχετική τροπολογία και από αυτού. Αυτά για την ώρα. Προσβλέπω στη συνέχεια των εργασιών μας. Ε, κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την κυρία Ντελβό και τους συνεργάτες της, γιατί πιστεύω ότι αυτή ήταν ε, μία από τις εκθέσεις που διαβάζει κανείς ευχάριστα. μπορεί κανείς, διαβάζοντας την έκθεση, να καταλάβει την ουσία. Από τις τροπολογίες που υποβάλαμε οι συνάδελφοι και εγώ, ίσως να υπάρχουν δύο ή τρία ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Το πρώτο έχει να κάνει με την νομική προσωπικότητα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί στις συναντήσεις μας μέχρι τώρα θα δώσουμε στα ρομπότ αυτή την νομική προσωπικότητα ή όχι. Και αν ναι, για τι σκοπό θα έχουν αυτή την νομική προσωπικότητα τα ρομπότ. Όπως φαίνεται και από τις τροπολογίες των συναδέρφων, θα υπάρχει ένα εύρος από το να μην προσφέρεται αυτή η νομική προσωπικότητα, ή από αρρωγή, για παρετέρω ανάλυση και άλλα. Το δεύτερο ζήτημα, σχετικά με το οποίο έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες, είναι η έκθεση αυτή, δίνοντας την νομική προσωπικότητα, πώς όλα αυτά συνάδουν με τα συστήματα ασφάλειας, τα φορολογικά συστήματα των χωρών μελών. Όπως είπε και ο προλαλής σας, τα ρομπότ σίγουρα θα έχουν κάποιες επιπτώσεις στη βιομηχανία μας, στην οικονομία μας τελικά. Κανείς δεν τον αμφισβητεί αυτό. Η δυσκολία όμως που αντιμετωπίζουμε έτσι είναι είμαστε εμείς ε, ε, σε θέση να πούμε τι συστήματα φορολογικά και κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καλύπτουν την περίπτωση αυτή. Ίσως χρειάζεται να το μελετήσουμε περισσότερα για να δούμε τι προτάσεις πρέπει να κάνουμε και να εξεταστούν βέβαια όλες οι νομικές πτυχές οι σχετικές με τα ρομπότ. Αυτά είναι τα δύο κύρια ζητήματα σχετικά με τα οποία έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες από πολλούς βουλευτές της ομάδας μου και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το τρίτο που είναι η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία η οποία σίγουρα θα έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για να βρίσκει λύσεις σε τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ντελβό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους και τα σχολιά τους. Συμφωνώ με την κυρία Κομοντίνη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Πρέπει να πω ότι είναι μια δουλειά που σίγουρα όλους μας ε, ενθουσιάζει και είναι και το θέμα του μέλλοντος. Εδώ δεν θέλουμε να μιλήσουμε φυσικά για science fiction, ούτε για θέατρο, ούτε μυθιστορήματα. Ναι, μ' αρέσει εμένα βεβαίως η επιστημονική φαντασία, μ' αρέσουν και τα μυθιστορήματα, ναι, αλλά στην έκθεση αυτή θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι θέμα του μέλλοντος και διαπιστώνουμε ότι τα ρομπότ ήδη βρίσκονται μεταξύ μας. Σίγουρα ο καθένας μας έχει συναντήσει κάποιο ρομπότ στον κύκλο του και ίσως χωρίς καν να συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ρομπότ. Ένας λοιπόν από τους στόχους της έκθεσης αυτής ήταν ακριβώς να προκαλέσει συζήτηση και να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση για το τι συμβαίνει γύρω μας τελικά. Γιατί διαπιστώνουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις πάνε πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μάλιστα φανταζόμουν όταν άρχισα να δουλεύω πριν από δύο χρόνια πάνω στα ρομπότ. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Τα drones είναι το δώρο που τα περσινά Χριστούγεννα προσφέρθηκε περισσότερο. Άρα δεν μιλάμε για ουτοπία. Από εκεί και πέρα χρέος μας και υποχρέωσή μας πιστεύω είναι να προκαλέσουμε τη συζήτηση και να είμαστε προσεκτικοί. Αν δεν θέλουμε τα πράγματα να προχωρήσουν χωρίς κανένα νομοθετικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τις αξίες μας αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η βιομηχανία μας είναι, καλή, έχει καλές επιδόσεις, αλλά ομολογώ αν είναι να ζήσω με ρομπότ, ε, ζήσω με ρομπότ ευρωπαϊκά και όχι η κινέζικα ή κορεάτικα. Αυτό λοιπόν που προτείνεται εδώ είναι δύο στάδια. Πρώτον, να δούμε τι πρέπει να ρυθμιστεί τώρα, αμέσως, και σίγουρα το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να λυθεί γρήγορα και γι' αυτό και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προτείνει ανακανονισμό, μια οδηγία και το πλεονέκτημα είναι ότι αν τώρα θέτουμε τις αρχές, αυτές θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή στις χώρες μέλη χωρίς να έχουν νομοθετήσει χώρες μέλη από μόνες τους και μετά εμείς να τρέχουμε από πίσω για να έχουμε εναρμόνιση της νομοθεσίας αυτής. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβλέψει τι γίνεται, να ενισχύσει την έρευνα, να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την έρευνα και όχι μόνο την έρευνα την τεχνολογική, αλλά και έρευνα επί των συνεπειών που τα ρομπότα αυτά θα μπορούσαν να είχαν στην καθημερινότητά μας και να μας προτείνει διάφορα σενάρια επ' αυτού. Γιατί εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της ρομποτικής στην απασχόληση. Θα έχει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να προετοιμαστούμε και να μελετήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Εξού και το ερώτημα θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε ένα νομικό καθεστώς στα ρομπότ. Εγώ δεν λέω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Λέω όμως ότι πρέπει να εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά, να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να βοηθήσει μια τέτοια νομική προσωπικότητα και σε τι θα συνίσταται ακριβώς. Πρέπει να φορολογούνται τα ρομπότ. Γιατί αν δεν έχουμε τέτοια έσοδα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την υγεία κλπ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα τεθούν βάσει σεναρίων που ελπίζουν να μην υλοποιηθούν. Αλλά αν ναι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η απασχόληση θα αλλάξει. Ότι η δεξιότητες, τα προσόντα τα οποία θα πετούνται μεθαύριο από τον κόσμο, από τους εργαζόμενους θα είναι διαφορετικά. Και άρα η πρόκληση για το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τεράστια. Πρέπει πάντα να υπενθυμίζουμε στην κοινή γνώμη ότι έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική αλλαγή της αλυσίδα παραγωγής και του κόσμου της εργασίας. Και άρα πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό είναι ο σκοπός. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι αυτός ο σκοπός. Δεν λέμε ότι θέλουμε την χη λύση για αύριο, λέμε όμως προσοχή. Γι' αυτό και προτείνουμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Γιατί βλέπουμε ότι άλλες ήπειροι δημιουργούν τέτοιες υπηρεσίες. Χρειάζονται, συνεπώς, ένα συνομιλητή και από εμά, ο οποίος να διαθέτει την πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται και να μπορεί να βοηθήσει για το θέμα της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, κλπ. Πρόσφατα το είδαμε με hackers που κατάφεραν να παραλύσουν ολόκληρα συστήματα. Και αυτό μέσω των στοιχείων που είναι διασυνδεμένα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε υψηλού επίπεδου ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε την έκκλησή μας. Σίγουρα είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να κάνει μόνο το Κοινοβούλιο, μπορούμε όμως να ζητήσουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Δεν θα επιμείνω περισσότερο, αλλά απλώς σας λέω ότι χαίρομαι πολύ που μπορώ να συνεργαστώ με τους συντονιστές, με τους σκιώδες συζητητές και βεβαίως με τους συζητητές των άλλων έξι κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση με ευρεία συνένεση, γιατί αν θέλουμε να περάσει το μήνυμά μας πρέπει να έχουμε και ευρεία πλειοψηφία, ώστε να αναλάβουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη, που είναι η εξέταση των τροπολογιών στην τήσια έκθεση για το 2014 όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Το λόγο έχει ο κύριος Καρύμου, εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για τις τροπολογίες τους στο σχέδιο αυτή. έκθεσης. Πολλές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενό μου και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε πρόοδο για τις διαπραγματεύσεις. Μπορώ να στηρίξω τις τροπολογίες των συναδέρφων που λένε ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι ε, μερικές από τις κύριες και όχι οι κύριες. Συμφωνώ ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα και οι σχετικές αποφάσεις δικαιολογούνται από την Επιτροπή, από διάφορα σώματα. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δίνει καλύτερη αιτιολόγηση όταν πρόκειται για αποφάσεις επικουρικότητας και αναλογικότητας. Τώρα, όσον αφορά το βαθμολόγιο αξιολόγησης, την αξιολόγηση για το 2014, 32% των αξιολογήσεων αντικτύπου καταλήγουν σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό, γιατί κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να το διαγράψουν αυτό, ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο πακέτο ρύθμισης για το 2015. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λογοδοτεί και να φροντίσουμε να γίνουν βελτιώσεις και να εφαρμόζονται αυτές και στους ελέγχους που γίνονται για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Τώρα για την ετήσια έκθεση, τις ετήσιες έκθεσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζω τις εκκλήσεις που κάνουν συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους για περισσότερες λεπτομέρειες και μια καλύτερη ανάλυση όσον αφορά την αναλογικότητα. Τώρα, θα ήθελα να κοιτάξουμε επίση λίγο περισσότερο τι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τις εκθέσει των Εθνικών Κοινοβουλίων για την διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλύπτουν και την επικορκότητα και την αναλογικότητα. Να το δω αυτό με τους σκιώδες εισηγητέ. Κάποιοι συνάδελφοι απέρριψαν την πρότασή μου για αιτιολογημένε γνωμοδοτήσει προκειμένου να περιλαμβάνονται αιτιολογήσει για την αναλογικότητα και αυτό να περάσει και στην επόμενη αναθεώρηση, άλλοι το στηρίζουν. Νομίζω ότι η αναλογικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ορισμένες υποχρεώσεις για λογοδοσία ήταν ε, κάπως ε, υπερβολικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επανεξετάζει είναι σημαντικό οι νομοθέτες να αναγνωρίσουν ότι η νομοθεσία μπορεί να είναι προβληματική για μικρές επιχειρήσεις και όταν συντάσσει ε, προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκέφτεται η υποχρέωση αυτή των επιχειρήσεων για να υποβάλουν εκθέσεις είναι κάτι αναλογικό ή όχι. Επίσης, κάποιοι συνάδελφοι, εξ αριστερών κυρίως, και αυτό με απογοήτευσε, δεν στηρίζουν την πρότασή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συστηματικά αξιολογήσεις για την αναλογικότητα για να εξετάζονται οι διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και να προτείνονται δράσεις όσον αφορά άτομα, επιχειρήσεις και μικρές και μεσές επιχειρήσεις κυρίως. Όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει καθοδήγηση από εμά για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η αναλογικότητα, δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν προβλήματα με την τρέχουσα νομοθεσία. Κατά τα άλλα, στηρίζω του συναδέρφου που τονίζουν το θέμα των ε, περιφερειακών κοινοβουλίων όσον αφορά την αναλογικότητα, αν και αυτό βέβαια ισχύει μόνο για μερικέ χώρε μέλη, όχι για όλε. Πολλοί συνάδελφοι έχουν υποβάλει και τροπολογίε στην πρότασή μου για την κόκκινη κάρτα και για το όριο για την κίτρινη κάρτα προκειμένου αυτό να αλλάξει. Με εκπλήσει αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα πλειοψηφία στην Επιτροπή μας για κόκκινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συζητήσουμε τα όρια για τα εθνικά κοινοβούλια που ακολουθούν τις διαδικασίες της κίτρινης ή της πορτοκαλή κάρτας. Για την πράσινη κάρτα τώρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Θα φροντίσουν να υπάρξει κάποιο συμβασμό, να στηρίξουν οι συνάδελφοι την ιδέα που νομίζω ότι ήδη τη στηρίζουν και αυτό με χαροποιεί. Έχω ετοιμάσει και κάποιο συμβασμό όσον αφορά την παράταση της προθεσμίας για τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να εκδίδει μια αιτιολογημένη γνώμη δεδομένου ότι είναι κάτι που έχουν ζητήσει πολλά εθνικά κοινοβούλια. Κάποιοι συνάδελφοι στηρίζουν την πρότασή μου για 12 εβδομάδες Ελπίζω ότι η πλειοψηφία των συναδέρφων θα μπορέσει να συμφωνήσει. Όσον αφορά την πρότασή μου για κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την επικουρικότητα και την αλογικότητα, θα κοιτάξω ποια θα είναι τελικά η διατύπωση από αυτού. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει μια μικρή αλλαγή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα τέλη Ιανουαρίου του 2017. Στο μεταξύ θα κυκλοφορήσω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και θα έχω και συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές εφόσον καταστεί αυτό αναγκαίο. Ευχαριστώ τους συναδέρφους για τη συνεργασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όλοι μαζί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Α, κύριε Αντελβό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρύμ για το έργο του. Τον ευχαριστώ επίσης και για τη συνεργασία του. Δεν συμφωνούμε όσον αφορά την επικουρικότητα, υπέβαλε όντως τροπολογίες. Και κατάλαβα ότι θέλετε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις. Όμως, ξεχνάμε μια αρχή της επικουρικότητας, γιατί η επικουρικότητα σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο και όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη. Συνεπώς εμείς εδώ συχνά συζητάμε ε, για τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται όσο γίνεται πιο κοντά στο πολίτη, αλλά αγνοούμε το θέμα της αποτελεσματικότητας της δράσης. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι στηρίζω, καταλαβαίνω να γίνονται ε, μελέτες αντικτύπου, τη σημασία τους, τη διαφάνεια, για να γνωρίζουμε ακριβώς πώς εφαρμόζονται αυτές οι αρχές, την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως, θέλω συγχρόνως να επενθυμίσω ότι έχουν γίνει πολλά, γιατί ολιγμένες γνώμες των Κοινοβουλίων έρχονται στην Επιτροπή μας. Ενημερωνόμαστε. Είδαμε και στην περίπτωση των αποσπασμένων ότι η προθεσμία που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι αρκετή, γιατί πήραμε πολλές τέτοιε γνώμες. Οπότε δεν νομίζω ότι η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους τα εθνικά κοινοβούλια αποτελεί εμπόδιο στο να παρέμβουν και να μας ενημερώσουν. Από την άλλη, μένα με απασχολεί το θέμα της αποτελεσματικότητας και έτσι εγώ προσωπικά νομίζω ότι είμαστε πολύ αργοί, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί πολύ, ότι οι διαδικασίες παίρνουν υπερβολικά πολύ χρόνο. Και δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι μια δράση είναι αναγκαία, να παρατείνουμε ακόμα περισσότερο τις προθεσμίες για να επιτρέψουμε άλλες διαδικασίες, άλλες μελέτες αντικτύπου και παράταση πάνω στην παράταση. Γι' αυτό θέλω να πω στον κύριο Καρύμ ότι είμαι έτοιμη και ευχαρίστως να συζητήσω μαζί του για να βρούμε λύσεις προς το συμφέρον μιας αποτελεσματικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος, δεν βλέπω να έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Ο κύριος Καρίμ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι ναι, είναι σαφέ για όλου του συναδέλφου, από όπου και αν προέρχονται, είτε συμφωνούν είτε όχι με την πρότασή μου, έχουν ε, μια προσέγγιση πολύ επικοδομητική και δραστηριοποιούνται. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για αυτή τη βοήθεια. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε περισσότερα από όσα διαφωνούμε. Και εκεί όπου διαφωνούμε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με συζήτηση να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στα σημεία 6 και 7 τώρα. Ανταλλαγή απόψεων για δύο θέματα. Διασυνοριακές ανταλλαγές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες όσον αφορά αντίγραφα κάποιων έργων που προστατεύονται από copyright. υπέρ των ατόμων τα οποία είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης ή για κάποιον άλλο λόγο δεν μπορούν να διαβάσουν τα έγγραφα αυτά, τα έργα αυτά. Ο κύριος Άντερσον είναι ο συγκητής. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης του Μαρακέσου για τους, που αφορά τους ε, τυφλούς και είναι μια συνθήκη η οποία αφορά την καλύτερη πρόσβαση σε βιβλία για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν ε, μειωμένη όραση. Ε, πρόκειται για την συμφωνία που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Διανοητική ε, και υπογράφηκε από 34 χώρες και έχει τεθεί σε ισχύ από το Σεπτέμβριο. Μέχρι στιγμής ε, ορισμένες χώρες δεν την έχουν επικυρώσει, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ε, θα γίνει σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχει επικυρώσει και κατά βάση πρόκειται για μια καλή πρόταση, μια θετική πρόταση. Είναι δύο καλές προτάσεις από την, της Επιτροπής. Είναι ισορροπημένες και πραγματικά είναι εφικτές εφαρμογές της συνθήκης του Μαρακές. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε πράγματι να τις υποστηρίξουμε. Πρόκειται για ένα πολύ ειδικό ε, θέμα. Γιατί έχει υπάρξει καθυστέρηση όσον αφορά, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την εφαρμογή αυτή τη συνθήκη και ελπίζω ότι με λίγη τύχη θα είμαστε σε θέση να διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Νομική Επιτροπή το Μάρτιο και ίσως με λίγο περισσότερη θα μπορούσαμε να το κάνουμε ακόμα και ε, νωρίτερα. Αλλά ο Μάρτιος ε, θεωρώ ότι είναι η ε, πιο πιθανή ημερομηνία. Επίσης θα ήθελα να πω ότι συζήτησα με την Επιτροπή όσον αφορά την διοργάνωση συναντήσεων για τους όσους ενδιαφέρονται να ενημερθούν περισσότερες σχέση με τις λεπτομέρειες των προτάσεων αυτών και ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια ημερομηνία για τέτοιου είδου ε, συναντήσεις ε, βάθο μελέτη. μελέτης. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντελβό. Αυτή τη φορά θα μιλήσω εξ ε, του συναδέλφου μας, του κυρίου Νεκρέσκου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί εδώ και θα διαβάσω αυτά που έγραψε. Ο Οργανισμός ε, Πνευματικής Ιδιοκτησίας διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και η συνθήκη του Μαρακές ε, ε, εγκρίθηκε το 24 Σεπτεμβρίου του 2013 και προβλέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά την κατοχήρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπέρ των τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση, με δυσκολίες πρόσβασης στα έντυπα μέσα. Αυτό αφορά συγκεκριμένα αντίγραφα βιβλίων ή άλλων εντύπων. Η εφαρμογή της συνθήκης θα επιφέρει πλεονεκτήματα για πολλά πρόσωπα τα οποία είναι τυφλά ή έχουν μειωμένη όραση όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε βιβλία ή έντυπα μέσα τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία. Τα ένα μέρη τη συνδίκη του ΜΕΣ θα παράσχουν κάποιε, διατάξεις, θα εκπονήσουν κάποιες διατάξεις σε ευθυγράμμιση με τη συνθήκη όσον αφορά για διασυνοριακά προσιτά αντίγραφα και εξασφαλίζοντας κάποιους περιορισμούς και εξαιρέσεις για ορισμένες ε, χώρες, τρίτες χώρες, αυξάνοντας τον ε, βαθμό πρόσβασης εκ μέρους των τυφλών σε βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα, ε, καθώς και οπτικοακουστικά προϊόντα. Η οδηγία λοιπόν θα ευθυγραμμίσει τον, την ενωσιακή νομοθεσία με τις διεθνείς δεσμεύσεις που προβλέπει η Επιτροπή του Μαρακέσου. Ο κύριος Νεγκρέσκου ε, πιστεύω ότι προσβλέπει με ζήλο να βρεθεί μια συμφωνία και πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι αναμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να επικυρώσει αυτή τη συνθήκη γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι δική μας υποχρέωση να επιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία υπογραφής της συνθήκης. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Άντερσον το εξή. Μπορούσατε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Το Μάρτιο είναι η απάντηση. Το Μάρτιο στην Επιτροπή Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι μάλλον το πιο ρεαλιστικό. Ε, το οποίο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά τυχεροί για να το πετύχουμε. Εάν εξασφαλιστούν οι μεταφράσεις, θα μπορούν να έχουμε την προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 7 Φεβρουαρίου και να γίνει η ψηφοφορία στις 22 ή στις 25 στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό αυτό το χρονοδιάγραμμα και θα μπορούσε πράγματι με κάποια τύχη, όπως είπα, να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντερσον για αυτή την πληροφορία. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το σημείο υπαριθμών 9 που αφορά το σχέδιο μιας γνωμοδότησης για τον συντονισμό συγκεκριμένων διατάξεων που εκπονήθηκαν ε, στις ε, ρυθμιστικές, στο επίπεδο ρυθμιστικών ή διοικητικών αρχών των χωρών μελών όσον αφορά τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες εν ώψη ραγδαία μεταβαλλόμενων μιας ραγδαία μεταλαμβαλόμενης πραγματικότητας ε, της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε εκμονήσει μια γνωμοδότηση και εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού υπάρχει μια γνωμοδότηση. Ε, είναι πολύ μακροτενής ο τίτλος αυτός. Πρόκειται για μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το, το Μάιο του 2016 διαθέτηκε ε, αυτή η πρόταση στο πλαίσιο της μιας στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ισορροπημένη πρόταση και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει και μια τεχνική πρόοδος, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά να ενισχυθούν και διάφοροι ε, παράγοντες ιδρώντες στην αγορά. Πρόκειται για έναν εξυγχρονισμό των οπτικοακουστικών μέσων στην αγορά, του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων, ε, πρόκειται για την τεχνολογική εξέλιξη στο πεδίο της τηλεόρασης των υπηρεσιών του διαδικτύου, καθώς και νέων ε, επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία εξελίσσονται εδώ. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογής, το οποίο μέχρι στιγμής ε, υπακούει στην, εμπίπτει στην οδηγία του 2010 και αφορά όλους τους παράγοντες στην αγορά των οπτικοκουστικών μέσων. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα προστασίας για την νεολαία και όσον αφορά την διαφήμιση. Κατά την τροποποίηση της οδηγίας δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι θα έχει ε, σημαντικές ε, επιπτώσεις σε πολιτιστικό επίπεδο και θα έχει και επιπτώσεις όσον αφορά την ε, πολυμορφία των μέσων καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης εκ μέρους των πολιτών. Σημαντικό είναι εδώ ότι η πρόταση αυτή για την τροποποίηση της οδηγίας λαμβάνει, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αφορά τα εξή ε, στοιχεία. Καταρχήν, την ε, διατήρηση της βασικής αρχής της χώρας προέλευσης γιατί ήδη έχει υποθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη προστασία των νέων και θα πρέπει να απαγορευθεί η ρητορική μίσους. Το ζητούμενο είναι επίσης οι αρμόδιες αρχές στον τομέα των επιτεκοακουστικών μέσων να γίνουν πιο ανεξάρτητες και να ενισχυθεί ο ρόλος τους. Η δική μας Επιτροπή διαδραματίζει εδώ ένα καθοριστικό ρόλο γιατί ασχολείται με διάφορα θέματα. Καταρχήν, πρόκειται για την ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και προστασίας των καταναλωτών. Ε, την καλύτερη ε, πρόσβαση στα περιεχόμενα των επιγραμμικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα για ένα, την εξασφάλιση ενός επαρκούς επίπεδου προστασίας για τους νέους ιδιαιτέρως όσον αφορά τα επιζήμια περιεχόμενα και την ρητορική μίσους που διαδίδεται μέσω του διαδικτύου. Πιστεύω ότι η δική μας Επιτροπή θα έπρεπε να ακολουθεί τον στόχο καταρχήν της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ε, δηλαδή οι δημιουργοί να έχουν ε, μία ικανοποιητική αμοιβή και θα πρέπει να εξασφαλίσει και τη δυνατότητα κάποιων επενδύσεων στον τομέα του πολιτισμού. Σας είπα επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη ανάληψη ευθύνης όσον αφορά την παροχή προστασίας στις ε, πλατφόρμες των βίντεο, να υπάρξει καλύτερη προστασία των δικημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να υπάρξει καλύτερη προστασία των νέων. Και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να δούμε ότι ε, υπάρχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης από τη μία. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να λειτουργεί ως πρόσχημα προκειμένου να απαγορεύονται τέτοιου είδους ε, πρακτικές. Δηλαδή στην πρόταση αυτή της ερωποποίησης θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε όλα αυτά να ανταποκρίνονται στις εθνικές διατάξεις και στο συνωσιακό δίκαιο και θα πρέπει ταυτόχρονα να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και παράλληλα να υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ε, διαφάνειας. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία και τη ε, ενδεχόμενη διεύρυνσή του, έχω την άποψή του ότι δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από έναν βασικό στόχο τη πρόταση τη Επιτροπή, δηλαδή ότι τα ε, υπηρεσίες, οι οπτικοχρηστικέ υπηρεσίε θα πρέπει ε, να υπάρξει μια προσέγγιση με τις επιγραμμικές υπηρεσίες. και μία προσέγγιση και σύγκληση με τους άλλους ε, τομείς του πολιτισμού. Τώρα, όσον αφορά τον χρονικό προγραμματισμό, 10 ε, Νοεμβρίου στι ε, στις 4 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ενώ η διενέργεια της ψηφορία στην Επιτροπή είναι στις 28 και 29 Νοεμβρίου ε, στην αρμόδια επί της ουσίας ε, επιτροπή, στην Επιτροπή Πολιτισμού, η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιανουάριο. Γι' αυτό ακριβώς τα όρια είναι κάπως, τα περιθώρια είναι κάπως στενά. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρεται. Κάποιος μας εκπλήσει, λέει, και δεν λοιπόν ενδιαφέρεται. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μονοπολίσω την Επιτροπή, θέλω να ευχαριστήσω την κύριο Νομίζω ότι χαιρετίζουμε όλη την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η αγορά των οπτικοκουστικών μέσων εξελίσσεται τάχιστα και διαπιστώνουμε σύγκληση μεταξύ τηλεόρασης και των υπηρεσιών των διαδικτυακών από το ίντερνετ. Πρέπει να εξυγχρονιστεί διόντως ε, η νομοθεσία. ομοιόμορφα να αντιμετωπίσουμε τους τομείς αυτούς. Χαιρετίζω το σεβασμό της αρχής εδαφικότητας, την πρόθεση των ευρωπαϊκών έργων, την προστασία του καταναλωτού βέβαια, που είναι κάτι που πάντα υποστηρίζουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, την προστασία των ανηλίκων και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της απαγόρευσης ε, των λόγων μυσαλλοδοξίας και ρατσιστικών ομιλιών και εκφράσεων που συναντούμε όλο και περισσότερο στα ΜΜΕ, που είναι κάτι ανησυχητικό. Και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, τον κατάλληλο, για να εμποδίσουμε τη διάδοση τέτοιων, τέτοιων μηνυμάτων. Ε, λοιπόν, οι διαφημίσεις και ανακοινώσει εμπορικού περιεχομένου, εγώ το μισώ αυτό που με διακόπτουν κάθε λίγο και λιγάκι οι διαφημίσεις. Δεν μπορώ να τι απαγορεύσουμε. Δεν μπορώ λοιπόν τέτοιου είδους τροπολογία να υποβάλω. Ε, η ενίσχυση του ρόλου της ομάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τα ΜΜΕ είναι κάτι καλό. Εντυπωσιάστηκα, θα έλεγα, από τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Λαμβάνοντας υπόψη νομοτής των άλλων επιτροπών για την έκθεση περί ρομποτικής θα πρέπει εδώ να επικεντρωθούμε επί των δικών μας αρμοδιοτήτων συντάσσοντας γνωμοδότηση. Διερωτώ με συνεπώς. Αυτή η διάδραση μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών φορέων εφόσον θέλουμε ελάχιστη εναρμόνιση μέσα της οδηγίας διατρέχουμε τον κίνδυνο κάτι να εγκρίνεται σε μια χώρα και να απαγορεύεται σε άλλη. Προβλέπει η οδηγία όμως ότι ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει μέτρα κατά μιας υπηρεσίας ακόμα και αν έχει έδρα σε άλλο κράτος μέλος. Έχω περισσότερο ερωτήσεις από ό,τι απαντήσεις. Μπορεί να μας διαφορετήσει ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τι αυτή περίπτωση με διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Τα κράτη-μέλη πώς θα διαθετήσουν τις διαφορές μεταξύ τους. Μήπως έχουμε πολλές συγκρούσεις μεταξύ εθνικών νομοθεσιών. Άλλο ερώτημα, η διαφάνεια. Στο άρθρο 2 θα το αλλάξουμε το κείμενο. Εκεί προβλέπεται κατάλογος παρόχων υπηρεσιών, οπτικοκουστικών υπηρεσιών, που είναι κάτι που αφορά την αρμοδιότητα του κάτω μέλους. Και λέει μετά το άρθρο, φροντίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ώστε οι ρυθμιστικέ, οι αρμόδιε ρυθμιστικέ αρχέ έχουν πρόσβαση στι ε, κατάλληλε πληροφορίε. Αυτό ο κατάλογο θα μπορεί να είναι δημόσιο. Σίγουρα δεν αποτελεί μυστικό. Έτσι κάθε ρυθμιστικό φορέα, αλλά και οι καταναλωτέ, θα έχουν πρόσβαση στον κατάλογο και θα μπορούν να γνωρίζουν ποιο είναι αρμόδιο, γιατί, για ποια υπηρεσία και σε ποιο κράτο μέλο. Αυτά είναι κάποια σχόλια. Ε, που απορρέουν. Με ενέπνευση οδηγία να προβώ τα σχόλια. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Άντρσον, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Ακόμα συντάσσω τις τροπολογίες μου, γι' αυτό θα είμαι λακωνικός. Αν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε κάτι για τις διαφημίσεις, κυρίως διαφημίσεις που έχουν σαν στόχο τα παιδιά, εάν υπάρχει δυνατότητα πρέπει κάτι να κάνουμε. Βασικό σημείο που με αφορά. Πρέπει να προσέξουμε, ούτως ώστε, να μην λάβουμε κάποια απόφαση επ' αυτού που αντιβαίνει την οδηγία περιεκτονικού εμπορίου, e-commerce. Δεν θα πρέπει να πιστέψουμε αυτό αυτό το χαρτοφυλάκιο να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο προς ενδιάμεση απόδοση ευθυνών. Μέσω ε, παραβίαση νομοθεσίας. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή την οδηγία θα πρέπει να τροποποιήσει. Να μην χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο σαν δούριο ύπο για να αλλάξει την οδηγία για την ε, ευθύνη των ενδιαμέσων. Αυτό είναι ένα τομέα επί του οποίου θα εστιάσουμε την προσοχή μα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπόη Αλόνσο έχει το λόγο. Συγγνώμη αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σα. Α, πολύ καλά, υπέροχα, υπέροχα. Από τι καλύτερε προφορέ που έχω ακούσει. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως συμφωνούμε μαζί σας και εμείς θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία που δεν είναι και εύκολη, ισορροπία μεταξύ προστασίας των ανηλίκων και των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων κυρίως της ελευθερίας της έκφρασης. Το εκτιμούμε ότι διαπιστώσατε ότι είναι δυσχερής η προσπάθεια. Συμφωνούμε λοιπόν μαζί σας. Κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς σας για να κατανοήσετε γιατί ακολουθήσαμε κάποια απορία, διότι προτείνεται να εισάγουμε μια τελογική σκέψη και, και δεν βλέπω να υπάρχει άθρο για αυτή την τελογική σκέψη. Αυτή η τελογική σκέψη που προτείνεται θα, θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες των ΜΜΕ να παρέχουν πληροφορίες περί περιεχομένου που θα μπορούσε να ε, είναι αρνητικό για τους ανηλίκους. Αυτό το, αυτή η λογική σκέψη συνοδεύει το άρθρο 6β που προβλέπει με νέα υποχρέωση. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το εξή. Θα πρέπει οι εκπέμποντες και οι πάροχοι ε, υπηρεσιών να δίνουν πληροφορίες στα προγράμματά τους αν υπάρχει βία, ναρκωτικά στο πρόγραμμα. Θα υπάρχει ένα μήνυμα που θα λέει προσέξτε, περιέχει το περιεχόμενο αφορά ναρκωτικά κλπ. Γιατί δεν προτείναμε να να μπει αυτή η υποχρέωση για πλατφόρμες κοινέ των ΜΜΕ, διότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Διότι η κοινή πλατφόρμα παράγει ε, ε, προϊόντα που ανεβαίνουν στο ίντερνετ και είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Στην πλατφόρμα Media Sharing Platform είναι δύσκολο να ελέγχει τα πάντα, όπως αν ανεβάσω εγώ ένα βίντεο και αυτή η media sharing platform να βάζει το σήμα ότι υπάρχει α, βία κλπ. Εγώ προβλέπω συγκεκριμένα άρθρα, συγκεκριμένε διατάξει και συμφωνώ με τον κύριο Άντερσον που συνάδουν με την οδηγία του ηλεκτρονικού εμπόριου. Θα υπάρχει ένα σύστημα ενημέρωση αν υπάρχει πρόβλημα με τα προγράμματα. Γι' αυτό δεν βάλαμε αυτή την ε, πρόβλεψη. Να απαντήσω τώρα στην κυρία Ντελβό. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα όταν υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες και άλλη χώρα προέλευση του προγράμματος, τη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ελάχιστη εναρμόνιση, αλλά ίσως κάποτε η χώρα που λαμβάνει ένα πρόγραμμα έχει αυστηρότερους κανόνες από τη χώρα από την οποία γίνεται έκπομπη. Και γι' αυτό έχουμε στο άρθρο 3 τη δυνατότητα παρέκκληση. Επιτρέπεται έτσι διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών για διευθυντή διαφορά. Να πούνε. ακούστε, κοιτάξτε, για μένα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε αυτό το μέτρο για την προστασία των ανηλίκων κλπ. είναι πολύ σημαντικό, κουβεντιάσουμε. Αυτό συμβαίνει και στι περισσότερε περιπτώσει διορθώνται τα προβλήματα. Σήμερα. Και πολύ συχνά ε, λέει εκείνο που εκπέμπει το πρόγραμμα θα προσαρμόσω το πρόγραμμα. Εκεί που δεν αν δεν δουλεύει το σύστημα αυτό παρεμβαίνουμε εμεί σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να βελτιώσουμε το μηχανισμό διευθετήσεω των διαφορών και η έργα να συμμετάσχει διότι έχει την τεχνογνωσία η ομάδα έργα, εφαρμόζουν την ε, οδηγία καθημερινά. Όπως είπατε κύριε Άντερσον, δεν βλέπετε γιατί αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τις γραμμικές υπηρεσίες. Για να εφαρμοστεί ο μηχανισμός εκεί της παρέκκλησης απαιτούνται τρεις παραβιάσεις. Αλλά όχι για ε, ε, υπηρεσίες κατά παραγγελία, on demand. Να σας εξηγήσω γιατί γίνεται διαφορά έχετε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα περιέχει λόγους μυσαλλοδοξίας. Οπότε εκεί υπάρχει παραβίαση. Αυτό συνέβη μια φορά. Αν υπάρξει άλλο πρόγραμμα, έχετε δεύτερη παράβαση. Άλλο ένα πρόγραμμα, τρίτη παραβίαση. Αν έχετε πλατφόρμα προγραμμάτων κατά παραγγελία video on demand, το πρόγραμμα είναι ακόμα συνεχές, συνεχώς παρόν και εξαρτάται το πόσες φορές χτυπάνε το πρόγραμμα και το ζητάνε οι πολίτες. Γι' αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να ζητήσουμε και να μετρήσουμε ότι θα γίνουν τρει παραβάσει. Και γι' αυτό δεν ζητάμε σε αυτή την περίπτωση τη παραβάση. Από τη στιγμή που υπάρχει μια παράβαση παραμένει μόνιμα και έχουν πρόσβαση οι πολίτε. Γι' αυτό το κάνουμε. Καταλαβαίνω την τροπολογία, αλλά αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο κάναμε τη διαφοροποίηση. Για τα υπόλοιπα Θα ήταν πολύ δύσκολο στο σύστημα παρεκκλήσεων, όπου ένα κράτος μέλος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν παραβάσεις και θα θέλαμε παρέκκληση όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση. Αν αυτή η κοινοποίηση είναι ατελής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει μια απόφαση. Είναι αδύνατον αυτό. Μιλάμε για μεθεμελιώδη ελευθερία. Μιλάμε για αναστολή θεμελιώδου ελευθερία και θεμελιώδου δικαιώματο ελευθερία τη έκφραση. Για να λάβουμε μια απόφαση με ατελή κοινοποίηση που προτείνετε εσείς είναι δυσχερέστατο. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και αν ζητούμε συμπλήρωση της κοινοποίηση είναι διότι έχουμε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Έχουμε λάβει κοινοποίησει ατελείς και δεν μπορούσαμε να λάβουμε απόφαση. Αν διορθωθεί και συμπληρώσει την κοινοποίηση το κάτω μέλο, μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε όμω αυτή η διαδικασία να επισημοποιηθεί, να θεσμοθετηθεί. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία το διαδικασία παράκαμψης της νομοθεσίας. Υπάρχει μια παρέκκληση από θεμελιώδη ελευθερία. Θέλουμε να υπάρχει διαβούλευση με την ομάδα έργα. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέω, αλλά προτείνεται ότι η έργα πρέπει να ετοιμάζει γνωμοδοτήσεις, αντί να υποβάλει γνωμοδοτήσεις. Δεν κατανοούμε. Πρέπει να υιοθετηθεί μια γνωμοδότηση. Έχει διαδικασίες η έργα, όπου υιοθετεί γνωμοθετήσεις γνωμοδοτή, συγγνώμη. Να προετοιμάζει γνωμοδοτήσει άνευ εγκρίσεως είναι κάτι που δεν κατανοούμε, ίσως κάτι δεν καταλάβαμε. Αυτά. Α, στην κυρία Ντελβό που πρότεινε κάτι. Δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την ενημέρωση, συμφωνούμε. Δεν το συμπεριλάβαμε στην πρότασή μας. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν ε, πράγματι, έχετε δίκιο, αν, αν είναι πιο ανοιχτή προσέγγιση και υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο εύκολη πρόσβαση πληροφορίες στις φυσικές αρχές, συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Καλώς. Καλώς. Τελειώσαμε με το σημείο αυτό. Με την άδειά σας, κύριε Σβιεύκα, ζήτησε το σημείο 12 να το εξετάσουμε τώρα για μια σύντομη ενημέρωση όσον αφορά την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να αλλάξει έτσι η μέρη στη διάταξη. Πρέπει να φύγω γιατί έχω μια άλλη συνάντηση. Θα επανέλθω όμως. Ναι, θέλω να σας ενημερώσω όσον αφορά την επίσκεψή μας στην Ελλάδα. Ο καθηγητής Χρυσόγονος ήταν μαζί μας. Ήταν μια αντιπροσωπεία ε, δύο μόνο. Και είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας στο μέλλον, γιατί ήταν λίγο περίεργο για να το πω έτσι. Μόνο δύο μέλη της Επιτροπής αυτής στην αποστολή αυτή στην Ελλάδα. Παρόλο που μας υποσχέθηκαν ότι θα ήταν πέντε τουλάχιστον και το πρόγραμμα είχε καθοριστεί με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά, είχε προετοιμαστεί για πέντε άτομα, ήταν πολύ γεμάτο και ομολογώ ότι ήταν μεγάλη απογοήτευση ότι τελικά συμμετείχαν τόσο λίγοι. Ο λόγος που έγινε η αποστολή αυτή ήταν οι αλλαγές στο ελληνικό νομικό σύστημα μετά την κρίση ή τώρα που η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, αν προτιμάτε. Θελήσαμε να διαπιστώσουμε η διασώμαση πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είχαμε λοιπόν ανταλλαγές απόψεων με καθηγητές και άλλους θεσμούς στην Ελλάδα. Είχαμε και το νέο αστικό κώδικα. Και μιλήσαμε και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον κώδικα αυτό και μιλήσαμε και με βουλευτές του, της Ελληνικής Βουλής. Πιο συγκεκριμένα, μιλήσαμε με δύο υποεπιτροπές στο ελληνικό, στην Ελληνική Βουλή. Συνερθήκαμε μαζί τους μέσα στη Βουλή. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Πολλές φορές οι προσεγγίσεις ήταν διαφορετικές. Είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον Είχαμε και μια ιδιαίτερα καρποφόρα συνάντηση με ένα νέο ελληνικό σώμα που είναι αυτό που επιθωρεί το κτηματολόγιο. Είναι ένα νέο σώμα. Πριν ήταν άγνωστο στο ελληνικό νομικό σύστημα, κάτι το οποίο εμένα με εξέπληξε. Γιατί ένα κτηματολόγιο για μένα, αν μη τι άλλο, είναι κάτι βασικό, το οποίο είναι αναγκαίο για να πολύ γη, ιδιοκτησία. Δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Μετά την Ελλάδα πήγαμε στην ε, Χαλκίδα. Και εκεί συναντηθήκαμε με δικαστές του τοπικού δικαστηρίου της πόλης δηλαδή. Ο καθηγητής Χρυσόγονος είχε ένα ραντεβού Μάλλον μια σημαντική διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, οπότε τελικά είχα την ευκαιρία τέτα τέτ να μιλήσω με τους δικαστές. Άκουσα για τις πιέσεις που έχουν την δουλειά τους, με ποιο τρόπο ασκείται η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου πώς ε, υπερισχύει ή όχι και η συζήτηση αυτή συνεχίστηκε και αργότερα με μια ένωση νομικών στη Χαλκίδα πάντα. Αύριο θα φιλοξενήσουμε εκπροσώπους του σώματος αυτού γιατί τους προσκάλεσα να έρθουν στην Επιτροπή μας, στη συνεδρίασή μας, για να δούνε πώς εμείς εργαζόμαστε εδώ και ποια είναι τα δικά μας θέματα. Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην άσκηση της δικαιοσύνης. Η ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τέτοιες ανταλλαγές δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που έχει κανείς βλέποντας τα πράγματα από μακριά. Τώρα αν εσείς θέλετε να σας δώσω κάποια λεπτομέρεια, να σας διαβάσω την έκθεση της αποστολής. Έχει πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάντως όλους και τη γραμματεία και όλους και να ακούσουμε και τον συνάδελφο βέβαια. Thank you, and uh, thank Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν στην Ελλάδα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη για όλους τους συμμετέχοντες. Λίγοι ήμασταν βέβαια. Είναι προφανές ότι υπάρχει σκεπτικισμό στην Ελλάδα όσον αφορά το νέο αυτό κώδικα, το που τέθηκε σε εφαρμογή πριν από μερικού μήνε. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα αρκετή εμπειρία, γιατί πρόσφατα εισήχθη στο νομικό μας σύστημα. Πάντως υπάρχει κριτική από ακαδημαϊκούς, από νομικούς και από δικαστές, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι κατά τη γνώμη μου τα προβλήματα της ελληνικής αστικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με μεταρρυθμίσεις του αστικού κώδικα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς δικηγόρους και πάνω από 40.000 είναι αυτοί για 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Ίσως η αναλογία αυτή να είναι η μεγαλύτερη κατακεφαλής ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι περισσότεροι δικηγόροι δημιουργούν τεράστιο φόρτο εργασίας για τα δικαστήρια. Ακόμα και αν ο αριθμός των δικαστών είναι υψηλός, που είναι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτό το φόρτο εργασίας μέσα σε λογικά χρονικά διαστήματα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν θα ήταν καλό να εξετάσουμε πιο αυστηρά τους δικηγόρους αυτούς οι οποίοι παίρνουν άδεια ώστε να περιοριστεί ο αριθμός τους σε ένα επίπεδο που να βρίσκεται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο. Και οι μεταρρυθμίσεις πάντα χρειάζονται χρόνο σε μια κοινωνία για να λειτουργήσουν. Αυτά, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσόγονο. Δεν βλέπω ερωτήσεις Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σιεύκα και να πάμε στο σημείο 10 που είναι σχέδιο γνωμοδότησης στην ε, έκθεση που έχει να κάνει με την εφαρμογή του κανονισμού 2004-113 για την ίση μεταχείριση αντρών και γυναικών στην ε, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η συγητής είναι ο κύριος Μαστάλκα, ο οποίος εδώ εκπροσωπείται από τον κύριο Χρυσόγονο, που αντικαθιστά τον εισηγητή. Έχετε το λόγο κύριε Χρυσόγονο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λείπει με αναρωτική ο κύριος Μαστάλγα και μου ζήτησε να παρουσιάσω εγώ την έκθεσή του αυτή για τον κανονισμό αυτό 2004-113 που εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η αρμόδια επί της επιτροπή είναι η Επιτροπή Γυναικών. Υπάρχει στον κανονισμό αυτό η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και υπηρεσίες. Λέει ο κ. Μαστάλκα ότι όλες οι χώρες μέλη έχουν πάρει μέτρα, αλλά ότι παραμένουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή. Ο κ. Μαστάλκα μεταξύ άλλων αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με την κατανόηση του τι είναι αγαθό και υπηρεσία. Ότι μερικές φορές δεν δίνεται αρκετά ξεκάθαρη αιτιολόγηση για τη διαφορά στη μεταχείριση ανδρών και γυναικών και δεν υπάρχει και επαρκή προστασία των γυναικών κατά τη μητρότητα και την εγκυμοσύνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με το περιεχόμενο και τι συνέπειε τη οδηγία. Στα συμπεράσματά του, ο συγητής ζητά από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες της οδηγίας και καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για την παρακολούθηση και να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες ε, δυναμικό της ε, οδηγίας, όπως ε, επίσης ο κ. Μαστάλκα θέλει ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και προσβλέπει στα σχόλιά τους. Κύριε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που όντως κάνει την προσπάθεια να έρθει σε επαφή και με τους σκιώδεις συγκητές για να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό κείμενο. Τα εξήγησε πολύ καλά ο κύριος ε, Χρυσόγονος. Όντως πρόκειται για την μεταφορά της οδηγίας αυτής του 2004 στην ένωμη τάξη των χωρών μελών όσον αφορά την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο σε μερικούς αλλά σε όλους. Να μην υπάρχει διάκριση λόγω φίλου. λοιπόν. Είτε πρόκειται για διάκριση, είτε πρόκειται για όχληση κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Υπάρχει το άρθρο 4.5 το οποίο δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι το πιο επίμαχο όταν φτάνουμε στην εφαρμογή γιατί είναι πολύ ασαφές και γενικό. Πάντως ο στόχος είναι προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι 28 χώρες μέλη έχουν μεταφέρει την ε, οδηγία στην νομοθεσία τους, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για την απασχόληση, αλλά όπως είπαμε πριν, για όλους τους τομείς της ζωής και στην εφαρμογή η οδηγία αυτή έχει κάποια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ πάντα τον εισηγητή και τον κύριο Μαστάλικα προσωπικά και σας. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Θα ήθελα να τονίσω μία συγκεκριμένη πτυχή, δηλαδή την ε, τυπική ε, ίση μεταχείριση των φύλων. Ε, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε εδώ να παραπλανηθούμε. Θα πρέπει να δούμε το θέμα ουσιαστικά. Θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση ε, ίσων των ίδιων υπηρεσιών. Γιατί υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει μία θετική ενδεχομένως ε, διάκριση υπέρ των γυναικών όσον αφορά το ζήτημα της μητρότητας. Πολλές ε, γυναίκες που γίνονται μητέρες διατρέχουν τον κίνδυνο ή να βρουν μια θέση εργασίας ή να απολέσουν την ε, θέση εργασίας που ήδη έχουν για να διατηρήσουν λοιπόν, προκειμένου να διατηρήσουν θέση εργασία τους, ορισμένες ε, παρετούνται από το δικαίωμα της μητρότητας και αυτό το φαινόμενο προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις σε ορισμένες χώρες. Και νομίζω ότι αυτό, σε αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να τεθεί ένα τέλος, λαμβάνοντας κάποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας θετικής διάκρισης των γυναικών, τα οποία να εφαρμοστούν και από τις επιχειρήσεις. Στην Πορτογαλία η μεγαλύτερη τράπεζα ε, επί πολλές δεκαετίες δεν προσελάμβανε καθόλου γυναίκες γιατί ε, θεωρούσε ότι θα μπορούσαν βεβαίως να αποκτήσουν παιδί αυτό ήταν μέχρι την αρχή του 20ου αιώνα. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό και νομίζω ότι οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις θα έπρεπε να υποχρεωθούν πραγματικά να λαμβάνουν κάποια προστατευτικά μέτρα υπέρ των γενικών, ούτως ώστε πραγματικά να υπάρχει μια ουσιαστική συμμεταχείριση των δύο φύλων. Δηλαδή να προβλέπονται δυνατότητες για τις γυναίκες, ούτως ώστε να μπορούν οι γυναίκες να ολοκληρώσουν ε, την προσωπικότητά τους ως εργαζόμενες και ως ε, γυναίκες, ως μητέρες, χωρίς να χρειάζεται να παρτιστούν από τη θέση εργασία τους. Και οι δημόσιες υπηρεσίες θα έπρεπε να δώσουν ένα θετικό παράδειγμα εδώ όσον αφορά την των δύο φύλων. Τα δικαστήρια στην Πορτογαλία τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια επί παραδείγματι έχουν ε, δικαστίνες, ε, γυναίκες εισαγγελείς, αλλά στο το στα νότατα δικαστήρια εκεί πραγματικά μπορεί να ψάξει τις γυναίκες με το φακό. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτή η συνταγματικά, ο συνταγματικ, η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ίσης των δύο φύλων να εφαρμοστεί ουσιαστικά στην πράξη. Θα πρέπει να γίνουν θετικά βήματα τους ώστε να τροποποιηθούν οι νομικές διατάξεις και να ευρεωθούν οι αρχές αυτές και στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος συνάδελφος που να θέλει να πάρει το λόγο, αλλά θα συνεχίσουμε με το σημείο υπαριθμών 11 που αφορά την ε, εξέταση των τροπολογιών όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση για τον έλεγχο του Μητρώου και τη σύνθεση των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Η συγκήτρια εδώ είναι η κυρία Κάουφμαν. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Έχουμε συνολικά 27 ε, τροπολογίες. Οι περισσότερες ε, από αυτές προέρχονται από τον κύριο Μπούντα, που πραγματικά βελτιώνουν το κείμενο και το καθιστούν πιο ισορροπημένο και επικεντρώνονται στα θέματα διαφάνειας και ιδιαίτερα στο θέμα της ισορροπίας ε, στην σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα μπορέσω να στείλω όλους τους συναδέλφους ε, τις προτάσεις ε, συμβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις συγκητές. Τρεις τροπολογίες, οι 25, 26 και 27 αφορούν την, ε, ε, τις ε, αιτιολογικές σκέψεις και την παράληψή τους. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να, υπάρξουν αυτές, να υπάρξει αιτιολογική έκθεση, άρα δεν μπορούν να γίνουν δεκτές αυτές οι τροπολογίες. Η δε... Νομίζω ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ούτως ώστε να μην προκύψουν προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να πάρει το λόγο. Α, ο κύριος Μπούντα, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο περιεχόμενο των ε, τροπολογιών σε σχέση με τον μηχανισμό στήριξης για τους εμπειρογνώμονες. Ορισμένοι συνάδελφοι κατέθεσαν κάποιες τροπολογίες εδώ, αλλά αυτό το οποίο ε, εννοείται εδώ ήταν η χρηματική στήριξη, χρηματοδοτική στήριξη. Βεβαίως μπορεί κανείς να ε, θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη υποστήριξη, όχι μόνο οικονομική. Ίσως θα μπορούσαν να το σκεφτούν οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να αφήσουμε τη δυνατότητα ανοιχτή να υπάρξει μια οικονομική αλλά και άλλη φύσεως υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κάφμαν. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πούντα. Πράγματι, ε, μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Εδώ, στο υπόβαθρο αυτού του θέματος ε, μιας ενδεχόμενης οικονομικής υποστήριξης, ε, αφορούσε τους εκπροσώπους των μικρών ε, μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίοι για την περίοδο αυτή ε, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις ε, υπηρεσίες τους και το να δούμε αυτό το ζήτημα μας οδήγησε στη σκέψη της δυνατότητας ενδεχόμενου μιας οικονομικής στήριξης. ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι οποίοι προσκαλούνται στις Επιτροπές Εμπειρογνώμων πράγματι να έχουν τη δυνατότητα να ε, συμμετέχουν χωρίς ε, διαφυγόντα κέρδη αν θέλετε. Τώρα έχουμε το τελευταίο σημείο, το 30, για το οποίο χρειαζόμαστε τον κύριο Χρυσόγονο. Uh, για να το κάνουμε κατά καταστροφές, ε, το σημείο 30. Ε, το ζήτημα της ασυλίας του κυρίου Πάξας έχει αναβληθεί. Ε, ας περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Χρυσόγονο, γιατί το σημείο αυτό το 30 δεν έχει αναβληθεί. Uh, Ωραία, λοιπόν, δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες ε, σχετικά. Θα συνεδριάσουμε αύριο στις 10 και υπάρχει και μια συνάντηση των συντονιστών στις 9 πριν. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα.